δύο μεθοδολογικά σχόλια. Κύριε Ταβάρες, έχουμε καθυστερήσει ήδη και δεν μπορώ να δεχτώ άλλα σχόλια πάνω στο θέμα της ουσίας. Μόνο διαδικαστικές παρεμβάσεις μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο λοιπόν. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα στη δήλωση του Συμβουλίου και, το, και της Επιτροπής σε σχέση με τις κλητεύσεις από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνω το λόγο στην κυρία Γιώρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Επίτροπε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο εκπροσωπεί τις αξίες και τις αρχές των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, Ευρωπαίων πολιτών όταν αναφέρεται στη συλλογή στοιχείων από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από εταιρείε ε, δημοσιότητες σε σχέση με το, τα λεγόμενα Wikileaks, σε σχέση με τις διαρροές εγγράφων. Το Συμβούλιο συμμερίζεται τι ανησυχίε του Κοινοβουλίου, αλλά δεν έχουμε πληροφορίε επί τη βάση των οποίων θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι οι Αμερικανικέ νομικέ ενέργειες έχουν παραβιάσει την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με την περίπτωση Wikileaks που αναφέραν οι κύριοι βουλευτέ, ο Γενικό ε, Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ποινική δίωξη για τα θέματα αυτά στι Ηνωμένε Πολιτείε και οι εισαγγελεί των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησαν να έχουν μια απόφαση δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να υπάρξει κλήτευση για την παράδοση δεδομένων προς αυτούς. Αλλά το Συμβούλιο δεν μπορεί να σχολιάσει αποφάσεις των δικαστικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών και εξάλλου δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες σε σχέση που θα μας βοηθούσαν να αξιολογήσουμε την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Υπήρξαν περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Twitter ε, πήρε το δικαίωμα από τα δικαστήρια να πληροφορήσει τους πελάτες της σε σχέση με αυτή την δικαστική απόφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις άλλων χωρών και σε περίπτωση ενός καταγγελό, μιας καταγγελόμενης αδικοπραξίας θα πρέπει τα οι άλλες χώρες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες. Είναι διαφορετικές οι διαδικασίες στις ΗΠΑ από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στις ΗΠΑ το δικαίωμα της κλήτευσης είναι ευρύτερο από ό,τι θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή διαδικασία δίωξης. Αυτό οφείλεται στην ε, νομολογία και την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι ένα θέμα λοιπόν για το οποίο το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κάνει σχόλια. Θα πρέπει να τύχουν σεβασμού οι κανόνες προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι και ευθύνη των εθνικών αρχών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εξασφαλίσουν το σεβασμό <clears throat> των κανόνων για τα προσωπικά στοιχεία και είναι στη δική τους αρμοδιότητα να εξετάσουν το κατά πόσο τα δικαστήρια τρίτων χωρών έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό δεν είναι ένα θέμα πολιτικής κρίσης για, για θέματα τα οποία έχουν χαρακτήρα subjudice και έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανικές αρχές στο παρελθόν έχουν προσπαθήσει να αποκτήσουν στοιχεία για πολίτες, των, ε, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν ε, Αποθηκεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επρόκειτο για στοιχεία που αφορούσαν τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών. Υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και κατέληξε αυτό σε, το 2007 σε μια συμφωνία και αυτή η συμφωνία θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί όπως ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η μεταφορά ε, χρηματοοικονομικών στοιχείων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ανείχνευσης τρομοκρατών της, των Ηνωμένων Πολιτειών και εδώ πάλι υπήρξε μία συμφωνία η οποία ανεκρίθη από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2010. Η περίπτωση του Twitter έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από ότι η περίπτωση του PNR των στοιχείων των επιβατών. Στην ε, προηγούμενη περίπτωση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας οι αρχές των ΗΠΑ συνέλεγαν ε, επιμακρών στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση του Twitter πρόκειται για μια συγκεκριμένη μονάχα διαδικασία ανάκρισης και έρευνας και θα πρέπει οι δικαστικές αιτήσει χωρών, τρίτων χωρών να γίνουν σεβαστές εκτός αν υπάρχουν αποχρόντες λόγοι για να τις απορρίψουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, λέω. Ο πρόεδρος η κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η προστασία των στοιχείων είναι ένα σημαντικό θέμα και νομικά πολύπλοκο. Είναι αυτονόητο ότι το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων που είναι θεμελιώδες δικαίωμα ισχύει και για τα ηλεκτρονικά για στην επεξεργασία δεδομένων. Ε, υπάρχουν και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, μάλλον, όπως και άλλα ε, δικαιώματα, μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να ορίζονται από τον νόμο και να είναι αναλογικοί και να δικαιολογούνται από θεμητά συμφέροντα, εθνική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, πρόληψη του εγκλήματος, προστασία της υγείας κλπ. Με βάση το, το νόμο, η σαπίνα, η κλήτευση είναι ένας νόμος που υποχρεώνει ένα άτομο να παρουσιαστεί σε μια συγκεκριμένη αρχή και να δώσει ορισμένε πληροφορίες. Η νομιμότητα μιας πράξης ορίζεται με βάση τον νόμο της χώρας όπου διεπράχθη το αδίκημα. Γι' αυτό η εκτίμηση της νομιμότητας, της ε, αναλογικότητας των ετοιμάτων των ΗΠΑ θα πρέπει να στηρίζεται στο Σύνταγμα των ΗΠΑ και το νομικό της σύστημα. Η Κομισιόν δεν έχει αρμοδιότητα για το πώς μια τρίτη χώρα εφαρμόζει τις δικαστικές της διαδικασίες σε ανακρίσεις σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες. Όταν Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν το Twitter εξέφρασαν τον προβληματισμό τους όσον αφορά την πολιτική και τον ιδιωτικό χώρο του Twitter. Ε, περιγράφεται αυτό όσον αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένου όταν χρειάζεται προκειμένου να συμμορφωθούν με νόμο ή νομοθεσία ή νομικό αίτημα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Επιπλέον, επειδή τα προσωπικά δεδομένα ε, ε, ζητήθηκαν μέσα στα πλαίσια ανακρίσεων σε σχέση με εγκληματικέ πράξεις η νομοθεσία προστασίας των δεδομένων των Twitter στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει. Η οδηγία της Ένωσης προστασίας δεδομένων δεν ισχύει για θέματα ποινικού δικαίου. Ούτε μια οδηγία πλαίσια σε θέματα συνεργασίας αστυνομίας και δικαστικών αρχών ισχύει στην περίπτωση αυτή, διότι καμία αρχή κράτους μέρους δεν ε, ε, είναι αρμόδια για να εκτελέσει τη δικαστική αυτή εντολή των ΗΠΑ και προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται από αρμόδιες αρχές από κάποιο κράτος μέλος. Συνεπώς, αυτά λέει ο νόμος. Ωστόσο, η παγκόσμια διάσταση της επεξεργασίας των δεδομένων δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειωθεί η προστασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μάλιστα, σε μια τέτοια διαδικασία παγκόσμιο επίπεδο ε, επιβάλλεται προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των δεδομένων των ατόμων και να διευκρινιστούν οι κανόνες, ιδιαίτερα σήμερα που όλο και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται σε αυτό που λέμε σύννεφο, κυβερνοσύννεφο. Τι θα κάνουμε τώρα σε σχέση με αυτά. Πρώτον, η πρόταση της Κομισιόν για μεταρρύθμιση της, του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων ειδικά θα εστιαστεί στις συγκεκριμένε αυτές προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών και της παγκοσμιοποίησης. Ιδιαίτερα όταν τρίτες χώρες, μάλλον παράγοντες σε τρίτες χώρες, έχουν σαν στόχο καταναλωτές της Ένωσης. Δεύτερο, ξέρετε ότι το Συμβούλιο 3 Δεκεμβρίου έδωσε εντολή στην Κομισιόν με στόχους μια διαπραγματευτική τη μελλοντική συμφωνία προστασίας δεδομένων με τις ΗΠΑ σε θέματα αστυνομίας και δικαστικής συνεργασίας. Ένας από τους κύριους στόχους της διαπραγματεύσης είναι να έχουμε δικαιώματα προστασίας των δεδομένων για άτομα από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού άσχετα με την εθνικότητά τους και διοικητική και δικαστική δυνατότητα προσφυγής και υπολογίζω στο Ευρωκοινοβούλιο να μας βοηθήσει σε αυτό. Βέβαια θα με ρωτήσετε στο μεταξύ τι κάνουμε πριν έχουμε στα χέρια μας αυτό το νέο εργαλείο. Συνιστώ ε, οι να είναι πάρα πολύ διαφανείς όσον αφορά τους ε, καταναλωτές, να τους λένε με σαφήνεια ότι οι υπηρεσίες τους διέπονται κυρίως από τον νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις ε, ανακρίσεις ποινικού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι καταναλωτές φεύγουν από την δικαιοδοσία της Ένωσης, ακόμα και αν οι ίδιοι δεν φεύγουν με το σώμα τους από την επικράτεια της Ένωσης. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Επίτροπε, τώρα οι σας. Ο κύριος Φως, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και το Συμβούλιο, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, εισηγήσεις τους. Πρόκειται για μια κλασική κατάσταση την οποία γνωρίζουμε στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο που ζούμε επί της αρχής. Φυσικά ε, σεβόμαστε το αμερικανικό δίκαιο και για τις δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζουμε με το παγκόσμιο μέσο του ίντερνετ προκύπτουν ε, προβλήματα. Αλλά ε, υπάρχουν και κάποιες κλασικές καταστάσεις όπου θα πρέπει για παράδειγμα να απαντήσουμε διοικητικά. Υπάρχουν θέματα ποινικού δικαίου σε ό,τι αφορά βάσεις δεδομένων. Και γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ με αυτά που είπατε Επίτροπε και εγώ αναρωτιέμαι για το πώς θα πρέπει να συνεχίσουμε να θα πρέπει να ρυθμίσουμε και να ανανεώσουμε τις βάσεις δεδομένων ή με αφορμή την κατάσταση αυτή να πούμε ότι θέλουμε να ρυθμιστεί ανάλογα η συμφωνία πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει η ανάγκη μεταφοράς δεδομένων σε ένα τέτοιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε φυσικά μια διαδικασία αυτή να μην επισκιάσει την επεξεργασία δεδομένων, αλλά καλό θα είναι να αναπτυχθεί η σωστή νομοθεσία, να συνεχιστεί η συμφωνία πλαίσιο και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ποινική δίωξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση δεδομένων, να φωτίσουμε το θέμα καλύτερα, σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επιτραπεί ή όχι η πρόσβαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε Φως, ο συνάδελφος Μωράης για δύο μισή λεπτά. Επίτροπε, νομίζω ότι είσαστε πολύ ικανοί και το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουμε στο μεταξύ. Γιατί είναι σαφές ότι είπα έχουν εκδώσει κάποιες κλητεύσεις κατά κοινωνικών δικτύων Yahoo, Twitter, Google αυτό δίνει πρόσβαση στη ΣΥΠΑ για τέτοιες ε, οντότητες όπως η Wikileaks και τρίτες οντότητες και φυσικά μιλάμε για Ευρωπαίους πολίτες, ε, αθώους πολίτες που είναι ε, με περίεργοι απλά νέοι άνθρωποι. Αυτοί θα πληχθούν ενδεχομένως από το καθεστώς αυτός. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και συνεχίζεται η κατάσταση Ασάντζ, αλλά αυτοί που πλήττονται ουσιαστικά από τις κλητεύσεις δεν είναι αυτοί που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την νομοθεσία τρίτων χωρών, αλλά θεωρώ ότι είναι νόμιμη και δικαιολογημένη η ανησυχία που επικρατεί στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να ε, εξηγήσουμε στον εκλογικό μας κοινό τι προστασία μπορεί να περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορούν ε, οι όροι αυτοί προστασίας να, αρούν, να αρθούν με μια κλήτευση απλά τον ήπα θα πρέπει να προστατευόνται οι πολίτες μας από υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκή νομοθεσία και ξέρω ότι προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεστε. Μέχρι τότε η οδηγία 9446 έχει προστατεύσει πολύ την αγορά αλλά έχει έρθει η ώρα να αναθεωρηθεί και να αυξηθεί το επίπεδο ασφαλείας. Θα διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με τη μελλοντική μας νομοθετική δουλειά. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θέλει να εισάγει η Επίτροπο στην αναθεώρηση προκειμένου να υπάρχει ευρωπαϊκή προστασία η οποία θα αντέχει στις ε, αμερικανικές κλητεύσεις. Να θυμόμαστε ότι δεν θα σταματήσουν τέτοια θέματα σε δίκτυα όπως το Twitter αλλά μπορεί να επισέλθουν και σε θέματα εθνικής επικυριαρχίας. Και αυτό αποτελεί μια ε, βασική ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Εν μέρει απαντήσατε ήδη σήμερα, αλλά νομίζω ότι είμαστε δικαιολογημένοι να είναι θεμητό να θέσουμε πιο πολλές ε, ερωτήσεις για πιο πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ και τώρα δύο λεπτά η κυρία Ιντφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και το Συμβούλιο, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με χαρά μου σημειώνω ότι συμφωνείτε με τις ανησυχίε μου. Να είμαστε σαφείς, δεν νομίζω ότι κανείς εδώ θεωρεί ότι είπα δρούσαν εκτός δικαιοδοσίας τους. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η δικαιοδοσία μέσα του διαδικτύου γίνεται τεράστια. Η δικαιοδοσία φαίνεται ότι επεκτείνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το πρόβλημα εδώ είναι το εξή. Παρά το γεγονό ότι οι εταιρείε που έχουν βάσει το διαδίκτυο, τι οποίε συζητούμε, κατά βάση έχουν έδρα στη ΣΥΠΑ, πολλοί χρήστε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το επιχείρημα το οποίο προβάλλεται από τους Αμερικανούς και από τα Αμερικανικά δικαστήρια και εδώ πέρα να σημειώσω ότι ήδη είναι παροχημένη αυτή η προφορική ερώτηση γιατί έχουν υπάρξει άλλες εξελίξεις. Τι λένε λοιπόν τα δικαστήρια ότι από τη στιγμή που κανείς χρησιμοποιεί το Twitter δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει οποιαδήποτε προσδοκία για ιδιωτική ζωή. Άρα οποιοδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει νομική προστασία πλέον, γιατί το Twitter έχει έδρα στις ΕΠΑ. Είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όπως είπε και η Επίτροπος Ρέντινγκ, στα πλαίσια της αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Λέτε ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιεί κανείς το Twitter συνενεί. Ε, μα τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συνένεση. Σημαίνει ότι είμαστε βγαίνουμε από τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάβουμε να έχουμε δικαιώματα νομικής προστασίας. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολλά να κάνουμε εδώ πέρα, αλλά να ρωτήσω τι προτίθενται να κάνουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προστατεύσουν νομικά τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα μιλήσετε στους ομολόγους μας, του Αμερικανούς, θα ζητήσετε πιο πολλές πληροφορίες, ίσως να υπάρχουν και άλλες εταιρείε που έχουν κλουτευτεί και αυτές. Και τέλος, είπατε Επίτροπε και κλείνω ότι δεν συγκρίνεται αυτή η υπόθεση με το SWIFT γιατί αφορά πολύ συγκεκριμένη έρευνα. Όντως, αλλά εκ παραλλήλου ζήτησαν και κλείνει το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ κυρία Ιντ. Φέρετε ο κύριο Άλμπρεχτ για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι αυτή είναι μία περίπτωση από πολλές. Έχουμε διαφορετική νομική κουλτούρα από τη μία όχθη του Αθλαντικού σε σχέση με την άλλη, ιδίω σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα και ιδιαιτερότερα όταν πρόκειται για αστυνομικά θέματα ή δικαστικά θέματα. Εγώ κλονίζομαι από την απάντηση που έδωσε το Συμβούλιο ότι είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με την ε, επικράτεια των ΗΠΑ και τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και επομένως δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο για τον νομικό χώρο προστασίας τη Ευρώπη. Εγώ το βρίσκω αυτό λαθασμένο. Εγώ το νομίζω ότι οι πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση το βλέπουν τελείως διαφορετικά το θέμα αυτό. Εμείς συνεργαζόμαστε σε διεθνέ επίπεδο όλο και περισσότερο με τις τι Πολιτείες σε θέματα αστυνομικά και σε θέματα δικαστικά. Και σήμερα όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε τη δικαιακή τάξη άλλων τρίτων κρατών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλε περιπτώσει, αλλά όλο και περισσότερο με τι ΗΠΑ όπου τίθενται θέματα προσωπικών δεδομένων. Και εγώ περιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο συγκεκριμένα, θα αναλάβει το θέμα αυτό και θα εξασφαλίσει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα να έχουν και εμπιστευτικότητα σε σχέση με το ίντερνετ, να έχουν προσωπικά δεδομένα για το ίντερνετ και να μπορούν να διατηρήσουν τις ελευθερίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε Άλμπρεχ. Ο συνάδελφος Στούπ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, το κόμμα για την ελευθερία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ε, προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων. Δεν είμαστε ε, κοντόφθαλμοι, είμαστε πραγματιστές. Θα πρέπει να ε, προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα του ανθρώπου, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τον ε, κίνδυνο της τρομοκρατίας. Γι' αυτό το σκοπό ε, όλοι παραχωρούμε ένα κομμάτι από την ιδιωτική μας σφαίρα. Οι χρήστες ε, του ίντερνετ και οι διευθύνσει IP για παράδειγμα θα πρέπει να προστατεύονται αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες τρομοκρατικών κινήτρων θα πρέπει να ε, υπάρχει δράση. Αν υπάρχει υποψία ε, στη ΣΥΠΑ για τρομοκρατικές ε, κινήσεις θα πρέπει να μπορούν να έχουν τα στοιχεία αυτά. Να μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν τα ζητάνε για πλάκα. Έχουν κάποιον καλό λόγο που τα ζητούν. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φαντριστούπ. Και τώρα περνάμε στον συνάδελφο Λόπες Αγγιλάρ για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ που παρά το προκεχωρημένο της ώρας είναι παρούσα σε αυτή τη συζήτηση της Ολομέλειας εδώ στις Βρυξέλλες για να ακούσει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να την εμψυχώσω για τη δουλειά αυτή που πρέπει να κάνει, τον επακαθορισμό δηλαδή των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ιδίω ό,τι αφορά την ανακοίνωση τη Κομισιόν για την προστασία των δεδομένων που θα παρουσιάσετε. Πρέπει να πω ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να βάλουμε του δείκτε του ρολογιού ε, στη σωστή ώρα. Να έχουμε αφενό τα εργαλεία και τι τεχνολογίε τη επικοινωνία, αλλά επίση να σεβαστούμε και την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που μεταξύ αυτών είναι η ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση δεδομένων ε, που πλήττουν μια, ε, ή θίγουν μια προσωπικότητα, αλλά και με τη συγκατάθεση των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει, ε, πρέπει να σεβόμαστε και το διεθνέ δίκαιο, γιατί εδώ μιλάμε για διμερεί διαπραγματεύσει μεταξύ κράτων, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτε χώρε και δι τι ΕΕ εδώ. Είναι σαφέ το μήνυμα που πρέπει να δοθεί. Οι κατευθύνσει. <clears throat> οι γενικές κατευθύνσεις καθώς και η οδηγία θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Και αυτό και για να παρέχεται η απαραίτητη αστυνομική δικαστική συνεργασία με τις κλητεύσεις και όλες τις άλλες ε, εντολές ή διαταγές ε, που θα πρέπει να εκδίδονται αλλά και για να υπάρξει ακριβώς ενίσχυση αυτής της διαδικασίας ε, και της ε, συγκατάθεσης και της πρόσβασης για να ξέρουν οι υπήκοοι των χωρών της Ένωσης ποια στοιχεία τους μεταβιβάζονται σε τρίτες χώρες και επίσης επαναλαμβάνω έχουν το δικαίωμα ακύρωσης ή διόρθωσης των δεδομένων που θίγουν την ιδιωτική τους σφαίρα, την προσωπικότητά τους και τα οποία υποβάλλονται σε αυτή τη μηχανοργανωμένη διαδικασία προσωπικών δεδομένων και μπορούν να, επεξεργαστούν στο πλαίσιο, να τύχουν επεξεργασία στο πλαίσιο του δικτύου. Και θέλω να τονίσω, σε ό,τι αφορά του ανηλίκου, τα δικαιώματά του πρέπει να προστατεύσουμε. Υπάρχουν κάποιες, κάποιοι περιορισμοί. Παραδείγματο χάρη, παιδική εργασία που δεν πρέπει να υπάρχει ε, και ε, κάποια άλλα δικαιώματα ιδιαίτερα για του ανηλίκου θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και ταυτόχρονα επαναλαμβάνω να γίνεται σεβαστή η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Εμείς θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην όλη διαδικασία και τη διαδικασία για την επικαιροποίηση ε, των διαφόρων κατευθυντήριων γραμμών και της οδηγίας και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα εργαλεία για τη διμερή συνεργασία με τρίτες χώρες και μεταξύ αυτών κυρίως τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστούμε και τώρα ένα λεπτό συνάδελφος Μέλτσερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παλιά παροιμία ότι αγαπάμε το, την προδοσία αλλά όχι τον προδότη είναι εδώ πέρα ε, πολύ επίκαιρο. τα, οι υπηρεσίες που δίνουν τις πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως προδότης. Αυτές, το τι γίνεται με τις πληροφορίες αυτές και το τι, ε, το τι καταδικάστηκε η Twitter είναι γνωστή, γνωστό. Κατά πόσο τα δεδομένα αυτά να τα χρησιμοποιήθηκαν από, άλλα, από άλλες ιστοσελίδες θα πρέπει να το μάθουμε, δεν το ξέρουμε ακόμα. Τα ονόματα των χρηστών και η παροχή διευθύνσεων email, το γεγονός ότι δεν θεωρούνται αυτό ως ε, ε μη προστατευμένα προσωπικά δικαιώματα είναι ενδεικτικό. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. President, it Πέρασε ώρα που να μου μπουν αυτοί οι διευμηνείς ότι πρέπει να πάρω το λόγο. Θα ήθελα να σταθώ λίγο σαν πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάσταση εδώ οικονομική, μια διάσταση εσωτερικής αγοράς πέραν των πολύ σημαντικών θεμάτων που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Εγώ συντάσσω την έκθεση της Επιτροπής μου για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρέντινγκ για το πράσινο βιβλίο πάνω στο οποίο βασίζεται. Είναι ένα από τα πολύ φιλόδοξα θέματα στα οποία αναφέρεται. Λέγει η κυρία Ρέντινγκ ότι αν εγώ έχω σαν Ευρωπαίος πολίτης τα δεδομένα μου σε ένα σερβερ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχω τα ίδια δικαιώματα πάνω στα δεδομένα αυτά σαν να ήταν τα δεδομένα σε ένα σερβερ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φιλόδοξη πρόθεση αυτή, ελπίζω να πετύχουμε την προσπάθειά μας. Αν ζητάμε πραγματικά κάτι τέτοιο, οι υπόλοιπες χώρες θα ζητήσουν δικαιώματα αμοιβαιότητας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Χάμπορ. Κλείνει η διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και τώρα το την στην ε, Επιτροπή President. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημερίζομαι τις ε, θεμητές ανησυχίες του Κοινοβουλίου στα θέματα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Ευρωπαίων πολιτών. Και επειδή ακριβώς συμμερίζομαι τις ανησυχίες παρουσίασε και την πρώτη ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο μεταρρύθμιση της οδηγίας του 95 θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Για να ανταποκριθούμε στα θέματα που τίθενται και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σήμερα, για το οποίο δεν έχουμε νομική ερώτηση, ε, απάντηση ακόμη. Δεύτερο στοιχείο. Νομίζω ότι σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, ε, οι ειδήσει είναι καλές. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ο Λευκός Σίκος έλαβε, έκανε ένα αποφασιστικό βήμα ανακοινώνοντας στις 16 συγκεκριμένα Μαρτίου ότι προτίθεται να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για την κατάθεση ενός ε, νομοσχεδίου για τα θέματα προσωπικών δεδομένων και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα στις ΗΠΑ το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και τις δικές μας προσπάθειες για τη Γενική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για αστυνομικέ ε, επιχειρήσεις και για δικαστική συνεργασία. Ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Και βασίζομαι βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσει στις προσπάθειες αυτές καθώς και στη μεταρρύθμιση οδηγία 95. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους του Συμβουλίου έχει το λόγο η κυρία Γκέρι. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. το θέμα είναι ότι είναι υποσυζήτηση η υπόθεση αυτή και απλά θα πρέπει προς το παρόν τουλάχιστον να επιβάλλουμε το κοινοτικό κεκτημένο ως έχει. Ξέρετε ότι έχουμε υιοθετήσει στο Συμβούλιο τα συμπεράσματα γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε. Θα ήθελα εδώ να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχάς. Μαζί της ε, επιμένουμε στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να ενημερώσουμε το κοινό. Και δεύτερον να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Ελπίζω λοιπόν ε, να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόψη αυτές τις δύο, αυτά τα δύο μικρά αιτήματα τα οποία της απευθύνουμε. Τίθεται επίσης και το θέμα της ενημέρωσης της ισχύουσας νομοθεσίας, διότι απλά πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες τεχνολογικές αλλαγές και προόδους. Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τις προτάσεις της ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας έλθουν υποτίθεται τον Ιούνιο δεν έχουμε και πάρα πολλές δυνατότητες ε, ε, βέβαια από εκεί και πέρα γιατί δεν θα έχουμε παρά μόνο ένα μήνα μπροστά μας αλλά είμαι βέβαιος ότι και η επερχόμενη Πολωνική Προεδρία θα τα φέρει πέρας ε, με επιτυχία. Λοιπόν, νομίζω ότι η ελευθερία ενημέρωσης από τη μία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων από την άλλη θα προχωρήσουν με επιτυχία χέρι με χέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε με το σημείο αυτό λοιπόν και περνάμε στο επόμενο. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η προφορική ερώτηση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας σε σχέση με την ποιότητα των καυσίμων και ιδίω για Α, λάθος διαβάζω, λάθος θέμα διαβάζω.